Witam ήρθατε. Ας μην περιμένουμε άλλο. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε τώρα τους υπόλοιπους συναδέλφους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι φεύγουν σήμερα και για το Βιετνάμ. Επομένως θα ετοιμάζονται προφανώς και δεν μπορούν να έρθουν στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Αγαπητοί συναδελφοί, έχουμε ένα μόνο σημείο στη ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους Επιτροπής σχετικά με τις προοπτικές και το μέλλον της αγοράς ζάχαρης. Ξέρετε ότι από πέρυσι έχουν μειωθεί σημαντικά οι τιμές της ζάχαρης και οι εκπρόσωποι του κλάδου της ζάχαρης έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι θα επέλθουν και περαιτέρω μειώσεις ε, στις τιμές του προϊόντος το 2017. Τα μέλη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον τα μέλη της δικής μας Επιτροπής ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μια παρουσίαση για τις γενικότερες προοπτικές του κλάδου της ζάχαρης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ζανζάκα Ζαφχελό, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις αρωτρές γες από την DG Agri. Έχετε λοιπόν το λόγο, κύριε Ζαφχελό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας προτείνω να εξετάσουμε πώς έχει η κατάσταση της αγοράς ζάχαρης και να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Και θα ολοκληρώσω την παρουσίαση αυτή με τις ε, προοπτικές ε, που ε, έχουν υποβάλει στον Επίτροπο Χόγκαν οι εμπειρογνώμονες για τον τομέα της ζάχαρης. Όντως είναι δύσκολη η χρονιά αυτή για τον κλάδο της ζάχαρης και κατάλαβα για ποιο λόγο θελήσετε να συμπεριλάβετε το σημείο αυτό στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Η κατάσταση στην παγκόσμια αγορά είναι πολύ δεινή για πέμπτη συναπτή χρονιά έχουμε ένα πλεόνασμα της παραγωγής της ζάχαρης σε σχέση με την κατανάλωση του προϊόντος και έχουμε λοιπόν ένα απόθεμα το οποίο συσσωρεύεται και το οποίο επιβαρύνει την αγορά του προϊόντος και γι' αυτό το λόγο οδηγούμεθα σε πολύ χαμηλές τιμές, 320 ευρώ ανά τόνο λευκής ζάχαρης. Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου καλύτερη. Η συγκομιδή για το 2014 ήταν ιδιαίτερα πλενοσματική, 19,4 εκατομμύρια τόνοι. Δεν περιμέναμε με τίποτα να έχουμε τέτοια παραγωγή ζάχαρης για το 2014 και ουσιαστικά προέρχεται από τις εξαιρετικά ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες που είχαμε στην Ευρώπη. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τώρα την παραγωγή αυτή με τις ποσοστώσεις παραγωγής που έχουμε θέσει, 6,5 εκατομμύρια τόνοι, καταλαβαίνετε ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει ε, να βρούνε πώς θα καταφέρουν να διοχετεύσουν αυτός επιπλέον 6,5 εκατομμύρια τόνους που περιβαίνουν ε, τις ποσοστώσεις παραγωγής. Αν δεν καταφέρουν να διοχετεύσουν αυτή την πλεονασματική ζάχαρη, τότε η ποσότητα αυτή της ζάχαρης θα πρέπει να περάσει στο επόμενο οικονομικό έτος. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε, επιβαρύνει ιδιαίτερα την αγορά ζάχαρης, διότι υπάρχουν, όπως βλέπετε, 2,5 εκατομμύρια τόνοι πλεονασματικοί, οι οποίοι θα πρέπει να μεταφερθούν στην επόμενη οικονομική περίοδο. Και αυτό με τη σειρά του έχει οδηγήσει τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στα πιο χαμηλά επίπεδα που είχαμε ποτέ από τη δεκαετία του 80, η τελευταία γνωστή τιμή αυτή του Απριλίου, δηλαδή 2015, είναι 417 ευρώ τόνο. Επιπλέον 200 ευρώ σε σχέση δηλαδή με την παγκόσμια τιμή που έχουμε. Οι παραγωγή ζαχαρότευτλων αντέδρασαν σε αυτή την πλονασματική παραγωγή και άρχισαν να μειώνουν τις ε, καλλιεργήσιμες εκτάσεις ζαχαρότευτλων κατά 15%. Καταλαβαίνετε ότι ε, το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο, γιατί αν κάνουμε μια προβολή σε σχέση με την παραγωγή, συνειδητοποιούμε ότι η παραγωγή μπορεί να μειωθεί κατά 3 εκατομμύρια τόνους και θα σταθροποιηθεί περίπου στους, στα 16 εκατομμύρια τόνους. Η κατανάλωση τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερή, περίπου δηλαδή στα 17 εκατομμύρια τόνους, Πράγμα το οποίο, παραδόξως, μολονότι είχαμε αυτή την ιδιαίτερα υψηλή συγκομιδή, όπως σας είπα, μας αναγκάζει να εισάγουμε, να εισάγουμε για να καταφέρουμε να αντισταθμίσουμε την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις ποσοστώσεις του 13,5, των 13,5 εκατομμυρίων τόνων και την κατανάλωση των 16,5 εκατομμυρίων τόνων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν καταφέρνουμε να έχουμε τις αναμενόμενες εισαγωγές. Και γι' αυτό το λόγο τα αποθέματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται και το, στο τέλος της περίοδου αυτής το απόθεμα δεν θα είναι υψηλότερο από ένα εκατομμύριο τόνους, δηλαδή είναι από τα χαμηλότερα αποθέματα που είχαμε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία του κλάδου της ζάχαρης. Δεδομένου λοιπόν αυτών των συνθηκών, δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για ιδιωτικά αποθέματα ζάχαρης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αναφερόμαστε καν στο ζήτημα αυτό, μια προσπάθεια περαιτέρω αποθήκευση ζάχαρης. Ανταυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σύντομα προτίθεται να εγκρίνει την πρώτη φάση εισαγωγών ζάχαρης για την περίοδο 2015-2016. Η Επιτροπή λοιπόν Ζάχαρης θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα και θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω, υπέρ της πρώτης αυτής φάσης εξαγωγών 650.000 τόνων προκειμένου να καταφέρουμε ήδη από την 1η Οκτωβρίου 2015 να ξεκινήσουμε τις πρώτες εξαγωγές. Όσον αφορά τώρα τις μελλοντικέ προοπτικές για τον κλάδο της ζάχαρης, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο αυτό, ιδίως όσον αφορά τις εξελίξεις που είχαμε από το 2006 και μετά διότι τα τελευταία 40 χρόνια δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αλλαγή όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ζάχαρη και παρόλα αυτά το 2006 είχαμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που κάλυψε την περίοδο 2006 με 2010. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης αυτής Μάλλον η μεταρρύθμιση αυτή εντάσσεται πλήρως στην γενικότερη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ξέρετε ότι ο, Ματσ, ο Επίτροπος Ματσαθλή, ο Επίτροπος Φίσλερ είχαν ήδη ξεκινήσει την ε, μεταρρύθμιση αυτή. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μεταρρυθμίζοντας τις ποσοστώσεις θα καταφέρναμε να, να καλύψουμε όλους τους τομείς γεωργικής παραγωγής και το μέση ζάχαρης είναι ο τελευταίος τομέας που καλύπτεται από τη μεταρρύθμιση αυτή. Έτσι λοιπόν όλοι μας οι εταίροι, οι εταίροι των χωρών ΑΚΕ αλλά και οι ίδιοι παραγωγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν μια πολύ μεγάλη περίοδο προσαρμογής η οποία επεκτάθηκε καθότι είπαμε ότι μόνο στο τέλος του 2017 θα σταματήσουν οι ποσοστώσεις παραγωγής. Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων αυτών έχουμε και ένα ταμείο 6 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αναδιαρθρωθεί ο κλάδος αυτός και προκειμένου ο κλάδος αυτός της ζάχαρης να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Ήταν ε, απόλυτο αναγκαίο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανοίξει πλέον πάρα πολύ τα σύνορά της στις εισαγωγές ζάχαρης από τις πιο φτωχές χώρες, από τις χώρες ΑΚΕ και στα πλαίσια πλέον του ε, ΠΟΕ δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε τις υψηλές εξαγωγές που είχαμε στο παρελθόν. Επομένως βρεθήκαμε αντιμέτωποι μια κατάσταση όπου όλο και αυξάνονταν οι εξαγωγές και όλο μειώνονταν οι δικές μας οι εξαγωγές. Χρειάστηκε λοιπόν να κάνουμε μια πολύ σημαντική αναδιάρθρωση γιατί περάσαμε από 183 εργοστάσια ζάχαρης τα οποία είχαμε πριν τη μεταρρύθμιση σε 102 τέτοια εργοστάσια και 4 επιπλέον εργοστάσια στη Ρουμανία και 3 επιπλέον εργοστάσια στην Κροατία. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια σημαντική μείωση της τάξης 40% όσον αφορά τη δυνατότητα παραγωγής μας. Και παράλληλα, ο κλάδος της ζάχαρης έχασε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Από 47.000 θέσεις εργασίας φτάσαμε στους 28.000 εργαζόμενους. Χάσαμε περίπου δηλαδή 20.000 θέσεις απασχόλησης σε αυτόν τον κλάδο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ο κλάδος της ζάχαρης χρειάστηκε να καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Παράλληλα, η διαδικασία επεξεργασίας ραφιναρίσματος εποφελήθηκε από την περίοδο αυτή για να αυξήσει την παραγωγικότητά του, τη δυνατότητα ραφιναρίσματος, η οποία αυξήθηκε από 2 εκατομμύρια σε 4 εκατομμύρια τόνους κοινέ αυτές δυνατότητες ραφιναρίσματος, επεξεργασίας αναπτύχθηκαν κυρίως στις γεωγραφικές εκείνες ζώνες που βρίσκονται μακριά από την παραγωγή ζαχαρότευτλων, δηλαδή ουσιαστικά στις περιφερειακές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, σας επενθυμίσουμε ότι η μείωση των θεσμικών τιμών από 632 σε 404 ευρώ ανατόνο μείωσε πολύ σημαντικά το παραδοσιακό χάσμα, την παραδοσιακή απόσταση που υπήρχε ανάμεσα στην, στην ευρωπαϊκή τιμή της ζάχαρης και την παγκόσμια τιμή της ζάχαρης. Ξέρω ότι πολλές φορές η ευρωπαϊκή τιμή ήταν τρεις φορές υψηλότερη από την τιμή της ζάχαρης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η μείωση αυτή της απόστασης, η μείωση αυτή της ψαλίδας ανάμεσα στις δύο τιμές κατέστησε λιγότερο ελκυστική την ευρωπαϊκή αγορά. Λιγότερο ελκυστική για τους ε, και για τους ε, ε, παράγοντες εκείνους που εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, σας είπα ότι ε, γίνανε κάποιες πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις από το 2006 και μετά, μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από το 2013 και μετά, και ουσιαστικά καταλήξαμε σε έναν κλάδο της ζάχαρης, ο οποίος είναι πλέον ανταγωνιστικός. Ε, θεωρούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πραγματικά τον ανταγωνιστικός αυτός ο κλάδος και ότι μπορεί πλέον να, αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις που προέκυψαν από το άνοιγμα των συνόρων αυτών προς τις πιο φτωχές χώρες, προς τις ναυτισσόμενες χώρες, προς τις χώρες ΑΚΕ, από τις οποίες λαμβάνουμε όλο και περισσότερες εισαγωγές. Τα δικαιώματα εισαγωγής διατηρήθηκαν και τις υπόλοιπες χώρες, τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν ανήκουν στις χώρες ΑΚΕ ή στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες. Από το 2009 όμως και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση βαθμιδών άρχισε να ανοίγει περισσότερο την αγορά της μέσω διμερών εμπορικών συμφωνιών με χώρες οι οποίοι είναι προμηθευτές ζάχαρης, όπως στην Κεντρική Αμερική ή με χώρες της Νοτίου Αμερικής, με την περιοχή των Άνθεων και με χώρες που είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ουκρανία, η Μολταβία, η Γεωργία. Και επίσης συνάφησαν και άλλες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, μάλλον πρόκειται να συναυτούν και άλλες ε, εμπορικές συμφωνίες, βρίσκονται την εξελίξη αυτή τη στιγμή, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, θα οριστικοποιηθούν σύντομα και θα τεθούν σε εφαρμογή. Άρα λοιπόν, με το τέλος των ποσοστώσεων και την απορρίθμιση που ακολουθεί, το γεγονός αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν μιλούμε για μια εξαφάνιση της Κομισιόν ή στην αγορά. Αντίθετα, η κοινή οργάνωση της αγοράς μένει ισχυρή. Παραμένει ισχυρή. Η βάση, το πλαίσιο της έχει αλλάξει. Και πλέον βασίζεται σε μια συμφωνία μεταξύ των καλλιεργητών και του βιομηχανικού κλάδου. Και μια δυνατότητα ο πλευράς κομισιών, εφόσον θα είναι απαραίτητο, να ενεργοποιήσει ιδιωτικά, αποθεματικά ή άλλα μέσα. Εξαγωγικές επιστροφές, εν πάση περιπτώσει παραμένουν κάποιες δυνατότητες. Αυτά λοιπόν Πρόεδρε τα μέτρα ε, συνιστούν ένα δίκτυο ασφαλείας πέραν του 17 και σε σχέση με την ομοθεσία πέραν του 17 έχουμε αυτή τη στιγμή σχέδια εν εξελίξη σχετικά ακριβώς με την ιδιωτική αποθυματοποίηση για το μέλλον και στην ομάδα που εξετάζει το σχέδιο αυτό το Κοινοβούλιο καλείται να αποστείλει εκπροσώπους. Τώρα έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα που κάνει η Κομισιόν για να προετοιμάσει το post 17 που είναι ακριβώς το αντικείμενο των, ε, της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Ομάδα η οποία ως στόχο έχει αφενός να συμβουλεύσει, να στηρίξει τον Επίτροπο Χόγκαν επί των μέτρων που θα πρέπει να αναλυφθούν και των διατάξεων που θα πρέπει να αποφασιστούν ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ενημέρωση και πληροφόρηση για τους ενδιαφερομένους φορείς ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες δυνατές οικονομικές αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε να βελτιώσουμε την ενημέρωση που διατίθεται στην αγορά, παρότι περιορίζεται αυτή η ενημέρωση από το γεγονός ότι υπάρχουν λίγες βιομηχανικές ομάδες, μερικές φορές ένας όμιλος ανακράτος, το οποίο μας αποτρέπει από μια λεπτομερέστατη ενημέρωση λόγω δεσμεύσεων εμπιστευτικότητος. Άλλη στόχευση της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι να εξετάσει τις ρυθμιστικές διατάξεις που θα πρέπει να μείνουν για την μετά τις ποσοστώσεις περίοδο. Δηλαδή το παρατηρητήριο τιμών θα πρέπει να διατηρηθεί ποια δεδομένα θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Κομισιόν με το στόχο δηλαδή του να έχουμε απόλυτη διαφάνεια ή στην αγορά. Μόλις ξεκινήσαμε τις συζητήσεις αυτές αλλά εξελίσσονται με μια κάποια συνένεση επί της αναγκαιότητας ε, να διατηρήσουμε το παρατηρείο τιμών και τις ε, κοινοποίησεις για τις τιμές και τα αποθέματα. Το κοινό λοιπόν καλείται, ξαναλέω, να αποστείλει αντιπροσωπεία. Τώρα, μετά το 17 θα έχει, θα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της αγοράς. Και οι δομές που πλέον θα είναι ανταγωνιστικότερες θα μπορέσουν να δώσουν όλη τους την αποδοτικότητα και δημιουργικότητα μαζί με την κατάργηση των εξαγωγικών περιορισμών πλέον, διότι καθότι δεν θα υπάρχουν ποσοστώσεις, δεν θα πρέπει να, δεν θα υπάρχει λόγος πλέον διακρίσεως και άρα θα έχει εκπνεύσει ο περιορισμός αυτός που υπήρχε ή στο παρελθόν. Εδώ θα υπάρξουν λοιπόν ευκαιρίες για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ζαχάρεως που οδηγούν σε κάποια στοιχεία αισιοδοξία εις ό,τι αφορά εις τους καλλιεργητές τους υπευθύνους ε, της επεξεργασίας ε, διογλυκόζης και την συνολική πρόσβαση σε μια αγορά χωρίς ποσοστώσεις και χωρίς τελωνιακές επιβαρύνσεις. Θα ήθελα με αυτήν την αισιόδοξη νότα κύριε Πρόεδρε να κλείσω Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο της Ερωικής Επιτροπής. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους ε, ε, των παραγωγών και της όλης αγοράς ε, ζαχαρέως στην Κροατία θα ήθελα να πω το εξή. Όπω είπε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν, οι τιμέ είναι χαμηλέ και εξακολουθούν να κατέρχονται από το 2004 χωρίς διακοπή. Και έχουμε φτάσει στα επίπεδα που έχουμε φτάσει σήμερα. Μιλούμε για μια συνολική μείωση του επίπεδου του 44%. Δεν πρόκειται για μια βιώσιμη κατάσταση στην Ευρώπη. Και είναι συνολικά ο κλάδος αλλά και οι μεμονωμένοι καλλιεργητές που υποφέρουν από την κατάσταση αυτή. Μιλούμε πλέον για 12 ευρώ τον τόνο και τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά σε περιπτώσεις κρίσεως κτλ. Αυτά όμως τα 162 εκατομμύρια ευρώ το έτος δεν χρησιμοποιούνται για τη ζάχαρη. Η άρση των ποσοστώσεων στη ζάχαρη θα εξακολουθήσει, θα συνεχίσει να οδηγεί σε προβλήματα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν κατά πόσον θα προχωρήσει η Κομισιόν αν έχει την πρόθεση να άρει τα μέσα αυτά ή αν για τους προϋπολογισμούς 16 και 17 θα χρησιμοποιηθούν τα μέσα αυτά ακριβώ για να βοηθηθεί ο τομέας της Δεχάρεως. Μαζί με την ε, πρώτη καλλιέργεια και την επεξεργασία, τη μεταποίηση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Ματί. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχάς ε, που αναλάβατε την πρωτοβουλία να εγγράψετε το θέμα αυτό σήμερα είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε πράγματι, μάλλον που έχουμε, μια ενημέρωση και παρουσίαση ο πλευράς ε, Κομισιόν για την αγορά της Ζαχαρίας. Εγώ άκουσα προσεκτικά την πληρέστατη αυτή παρουσίαση και σας ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι βασίζεται τα στοιχεία σας στην παραγωγή ζαχαροκαλάμου. Ζαχαροτέφτλου, με συγχωρείτε. Επομένως, ως προς τη διάκριση αυτή, ως προς την παραγωγή δηλαδή του ζαχαροκαλάμου και το μέλλον της, έχουμε μια σειρά ερωτήσεων. Να σας υποβάλουμε, ώστε να δούμε αυτή η ομάδα επιλογνωμόνων έχει λάβει υπόψη της την διάκριση αυτή, την παραγωγή ζαχαροκαλάμου και ποιες είναι οι υπεροπτικές εκεί συγκεκριμένα για τα μετά το 17. Και για να αντιληφθεί κανείς την διάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζομαι, να θυμίσω κάποια μεγέθη. Η παραγωγή ζαχαροκαλάμου δεν εκπροσωπεί παρά ε, ένα απειροελάχιστο ποσοστό της συνολικής παραγωγής της εβραϊκής δηλαδή περίπου 500 τόνοι το έτος 500.000 ε, τόνοι το έτος δηλαδή 3% της συνολικής παραγωγής και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που παράγει 66.000 66 μάλλον της 100 της συνολικής παραγωγής παράγει το 0,03% της συνολικής της παγκόσμιας δηλαδή παραγωγής. Γιατί το αναφέρω αυτό. Απλώς για να επιδείξω ότι με το 0,03% της παγκόσμιας παραγωγής είμαστε ενώπιον μιας απόλυτης αδυναμίας να επιφέρουμε, αν θέλετε, σημαντικές, ε, σημαντική επιρροή στην παγκόσμια αγορά. Και οδηγηθήκαμε στη μεταρρύθμιση αυτή που ξεκίνησε από το 2005 και που επιβεβαιώθηκε και πιο πρόσφατα. Δεν θέλω τώρα να κάνω σύνοψη ιστορική, αλλά θα ήθελα να καταλάβω εντός των συνθηκών αυτών πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Και θα ήθελα σε δύο επίπεδα να σας Υποβάλλω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς για τα ειδικά προϊόντα ζαχάρεως και τα οποία ανταγωνίζονται με τα προϊόντα ζαχάρεως που παράγονται από διάφορες χώρες που έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες μαζί μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ επιτρέψτε μου, εφόσον έχω τη χρονική δυνατότητα, να σας δώσω κάποια μεγέθη. Η αγορά της ειδικής ζαχαρέως είναι 250.000 τόνοι σε ευρωϊκό επίπεδο, δηλαδή λιγότερο του 1,5% της ευρωϊκής αγοράς. Και αυτή η αγορά είναι απολύτως ανοιχτή, όπως γνωρίζετε, στις τρίτες χώρες, στο επίπεδο του 50% για χώρες ε, ΑΚΕ και άλλες οι οποίες εισέρχονται χωρίς τελωνιακές δεσμαλογικές επιβαρύνσεις. Ο αντιγωνισμός αυτός είναι ζωηρότατος, εντονότατος, όλο και πιο έντονος μάλιστα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάβει να πολλαπλασιάζει συμφωνίες εμπορικών ελευθέρων συναλλαγών, μερικές τις διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή ακόμη, με χώρες που έχουν κόστη παραγωγής εξαιρετικά χαμηλά και με τις οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο εμείς να ανταγωνιστούμε ισότιμα με δίκαιους όρους. Και αναφέρομαι και στις ε, απόμακρες και περιφερειακές περιοχές της Ένωσης και υπερπόντιες. Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη, πραγματική ανάγκη, αυτά τα ειδικά προϊόντα ζαχάρεως να εξαιρεθούν των συμφωνιών ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών. Και σκέπτομαι τις μελλοντικές συμφωνίες με Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Ινδία, δεν θα τις αναφέρω όλες. Αλλά γνωρίζω ότι η Κομισιόν είναι μάλλον αρνητική σε μια ρήτρα ομαδικής εξαιρέσεως των ειδικών αυτών ζαχάρεων. Τώρα θα μπορούσε να υποβληθεί ίσως προς εξέταση ή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων το γιατί επί δεν μπορούμε να προτείνουμε μια διαφοροποίηση εντός του πλαισίου όλων των συμφωνιών ειδικά προϊόντα ζαχάρεως έτσι όπως θα το επιτρέπει η τελωνιακή νομοθεσία και διατάξεις και κατηγορίες. Και άλλο ένα να πω, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς καθότι επί των ποσοστώσεων που μιλούμε για τα ειδικά προϊόντα ζαχαρέως να προβλέψουμε να μην υπερβαίνουμε το 1,5% για το σύνολο των παραχωρήσεων που κάνουμε. Δηλαδή Εάν διαπραγματεύεται 10.000 τόνους η Κομισιόν, το διακύβευμα δεν θα ήταν για τα ειδικά προϊόντα ανώτερο των 100 με 150 τόνων. Ζητώ συγγνώμη για το τεχνικό της τοποθετήσεως, αλλά ήταν σημαντικό να υποθούν αυτά και να τα ακούσει η Κομισιόν για να μπορέσει να δεσμευτεί προς έναν τέτοιο προσανατολισμό, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την παραγωγή ζαχαροκαλάμου στις περιοχές μας και στην οποία έχουμε επενδύσει εκατομμύρια εκατομμυρίων. Σε διάφορα χρόνια έχουμε εξυγχρονίσει τα μέσα παραγωγής, έχουμε περί τα 30.000 άτομα που εξαρτώνται άμεσα από την αγορά αυτή, που είναι βασική εξαγωγική πηγή συγκεκριμένων περιφερειών και χωρών και εκεί θα έχουμε υψηλούς κινδύνους από την καταστροφή αυτής της παραγωγής. Όσο σε ό,τι αφορά τα προϊόντα επεξεργασμένης ζαχάρεως χίδιν, θα πρέπει νομίζω η Κομισιόν να σκεφτεί, να εξετάσει μέτρα τα οποία να είναι συμβατά και με τη μεταρρύθμιση αφενός αλλά και με την αντιστάθμιση των ε, συνεπειών για τους καλλιεργητές αφετέρου. Περιμένω τις απαντήσεις της Κομισιόν και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην μιλήσετε και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τότε θα χάσουμε την μπάλα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, λέει ο Νταντά. Εδώ πέρα μιλάμε βέβαια για το ζαχαροκάλαμο, γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκή επικράτεια. Θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε περισσότερο κατά καιρού. Εγώ θα μιλήσω για το σαχαρότεστιλο βεβαίω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση που πράγματι ήταν σχετικά σαφή. Όταν το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αποδεχθήκαμε την πολιτική βούληση Κομισιών και Συμβουλίου να φύγουμε από την πλαισιωμένη αγορά, από του συστήματος δηλαδή που υπήρχε ε, προηγουμένως από τη αυτά και μετά. Με τις ροές παραγωγής βλέπουμε ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι έχουμε φύγει από το καθεστώ των ποσοστώσεων ενώ ακόμα υπάρχουν. Ακούσαμε ε, στοιχεία για την παραγωγή 2014, δεν αναφέρθηκαν οι ποσότητες ζάχαρης ε, που ε, εισήχθησαν. Έχουμε πολλές διεθνείς συμφωνίες που σημαίνει ότι επιστρέφουμε καταργασμένη ζάχαρη χίβιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εισέχεται δηλαδή τέτοια καταργασμένη ζάχαρη, αλλά μήπως εισάγουμε περισσότερο από αυτό που προκύπτει με την αυστηρή του όρου από τις συμφωνίες. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το στάδιο καθεστώσεων των διαπραγματεύσεων συγγνώμη, μετά τις αποσωστώσεις. Ορισμένοι φορείς ε, προσπαθούν να προκλήσουν, προκαλέσουν την παρέμβαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για το άρθρο 101 της Συνθήκης. Θέλω να επενθυμίσουμε ότι στη διαπραγμάτευση της ΚΑΠ θέλαμε ε, να προβλέψουμε τι θα συμβεί μετά τις ε, ποσοστώσεις ε, στην αγορά γεωργικών προϊόντων και με πολύ συγκεκριμένους κανόνες για τον μεταγωνισμό. Επομένω, το Κοινοβούλιο θα μεριμνήσει ούτω ώστε η πολιτική συμφωνία που υιοθετήθηκε με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να γίνει σεβαστή από όλους τους φορείς και κανένα να μην προσπαθήσει να διεκδικήσει άλλες προτάσεις προς διαφορετική κατεύθυνση για την Κομισιόν. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ο Επίτροπος ε, έκανε συγκεκριμένε συστάσεις και παρατηρήσεις για τη διαφορετική μα μας θέση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ρεμπέγκα. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι σε χώρα την αγορά ζάχαρη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την λεπτομερέστατη ε, παρουσίαση και τα στατιστικά στοιχεία που μας έδωσε. Λέτε ότι η βιομηχανία έχει γίνει προβολικά ανταγωνιστική και γι' αυτό το λόγο τώρα χάνουμε θέσεις εργασίας και κλείνουμε εργοστάσια. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Πάνω πάνω από 180.000 άτομα απασχολούνται στον τομέα. Από το 2006 πάνω από 80 εργοστάσια έκλεισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 20.000 θέσει εργασία έχουν χαθεί, όπω τα λέγατε κι εσεί. Όταν καταργηθούν οι ποσοστό του 2017, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μία από τις πλέον απελευθερωμένες αγορές ε, ζάχαρης στον κόσμο σε άλλες ε, χώρες όπως η Ινδία, Βραζιλία, Ταϊλάνδη και αλλού ε, υπάρχει σαφή στήριξη του εθνικού κλάδου ζάχαρης. Εμείς λοιπόν πώς θα αντιδράσουμε, ποια θα είναι τα μέσα προστασίας των ε, καλλιεργητών μας. Τι ακριβώς έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το τομέα. Γιατί τα τελευταία δύο χρόνια με το καθεστώς των ποσοστώσεων βλέπουμε ότι ο κλάδος έχει συμβάλει στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Άνωσης ε, σε ύψους 320 ε, εκατομμυρίων ευρώ ε, εν είδη φόρων και το καθεξής. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε αυτόν τον κλάδο και την απασχόληση και τις επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο. Όλα αυτά συζητήθηκαν και στις 26 Ιανουαρίου στο Συμβούλιο Υπουργών και δημιουργήθηκε και μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα εξέταζε τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να μετριαστούν οι συνέπειες της κρίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επόμενη ε, συνεδρίαση αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, έχω τις εξής δύο προτάσεις. Να υπάρξει πολιτική συμμετοχή από πλευράς κρατών μελών στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και όχι μόνο ε, συμμετοχή τεχνοκρατών ε, των Υπουργείων, γιατί είναι και θέμα στρατηγικής πολιτικής. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών της ζάχαρης, δηλαδή του κλάδου της ζάχαρης, ε, δεν είναι ευπρόσδεκτη σε αυτή την ομάδα εμπρογνωμόνων. Όμως, έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν και να δουν την κρίση όπως τη βλέπουμε και εμείς. Και παρουσιάζουν ε, τα προβλήματά τους από πλευρά επενδυτών. Και θεωρώ ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δική τους γνώμη. Πρέπει να συμμετάσχει δηλαδή και ο κλάδος ε, σε αυτή τη συζήτηση. Τελευταία παρατήρηση. Εάν παραμείνει έτσι η κατάσταση, τα τελευταία τέσσερα εργοστάσια που παραμένουν στη Ρουμανία θα κλείσουν και θα πρέπει και εμεί να εισάγουμε ζάχαρη από άλλε χώρε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ήδη έχουμε υφιστάμενε υποδομέ και μετά θα πάμε να εισάγουμε ζάχαρη ενώ μπορούμε εμεί να την παράξουμε άνετα. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα χαθούν οι θέσει εργασία σε αυτόν τον κλάδο. ενώ προσπαθούμε να διαμορφώσουμε γενικά και να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Ευχαριστώ. Περιμένω να ακούσω και την ε, θέση τη Κομισιόν. Η ζάχαρη δεν είναι καλή για την υγεία όμως, ξέρετε. Δεν ε, με αναφέρετε, Πρόεδρε, αλλά ο γραμματέας με έδειξε. Εντάξει. Ήθελα τυπικά μόνο να πω ότι είμαι και εγώ καλλιεργητής ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό συγκεκριμένα εδώ. Ο καθένα μα αυτή τη στιγμή τώρα περιμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο να έρθει η προσφορά από την British Sugar, που είναι μονοπωλιακό όμιλο και θα είναι μάλλον άσχημα τα νέα, ε, μειωμένη ποσόστοση, μειωμένη τιμή. Ελπίζουμε να μας δώσουν μία τιμή που θα μας δίνει κάποιο ποσοστό κέρδους, παρότι ε, τα περιθώρια είναι στενά. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι και σε άλλα εμπορεύματα είναι χαμηλές τιμές. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος εύκολα να αλλάξει η καλλιέργεια και να πάει σε κάτι καλύτερο. Είναι πολύ άσχημη η χρονική συγκυρία. Ακριβώς επειδή έχει το μονοπόλιο, ελπίζουμε η British Sugar να ε, συμπεριφερθεί υπεύθυνα. Τώρα, εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε δύο δηλώσεις. Είπε ότι υπάρχει μεταφορά 2,5 εκατομμυρίων τόνων και μετά είπε ότι δεν υπάρχει πλεόνασμα ζάχαρης να αποθηκευθεί. Αυτό, μετά είπε ότι αυτό δεν έχει πολύ νόημα, δεν είναι λίγο αντίφαση και εγώ συμφωνώ. Μπορείτε λίγο να μας τα εξηγήσετε. Είτε υπάρχει πλεόνασμα είτε δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν εγώ δεν κατάλαβα καλά. Υπάρχουν ε, ευρωβουλευτές από τη Φιλανδία εδώ, δεν ξέρω ήταν μια χώρα που είχε τη δυνατότητα να μεταρρυθμίσει τον κλάδο της και να λάβει ε, επιδοτήσεις ε, που κατέστρεψε τη βιομηχανία της. Θα υπάρξει τώρα ζήτημα. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε κάτι να μας πει για τη Φιλανδία, γιατί δεν βλέπω πώς ε, μπορεί να συνεχίσουν εκεί τα πράγματα. Αναφερθήκατε στην περίοδο μετά το 2017 όταν θα καταργηθούν όλες οι ποσοστώσεις. Μπορεί να έρθει η καταστροφή. Και αν υπήρχε τον να αξιοποιήσουμε συγκεκριμένου ε, δείκτε, αυτή ήταν η ευκαιρία μα. Δυστυχώ όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τα πράγματα με το λεγόμενο MIFID, που θα κάνει τι ε, αγορέ αυτέ πολύ πιο δύσχριστες. Δεν θέλω τώρα να σας επικρίνω συνεχώς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί παρέχεται και κάποιες εφέλιμες υπηρεσίες όπως είναι το παρατηρητήριο τιμών για το γάλα και για τη ζάχαρη. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωφέλιμη υπηρεσία αυτή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξέρουμε ε, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Γιατί γι' αυτό τους πληρώνουμε εξάλλου. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω τη μαγιά και τους παραγωγούς ε, μαγιάς ε, για να υπάρχει διαφάνεια σε αυτή την αγορά μετά το 2017. Θα ήθελα λοιπόν να αξιολογήσουμε τις δύο αγορές ζάχαρης αντί για τη μία, όπου, δηλαδή η, η, η αγορά όπου χρησιμοποιείται άμεσα η ε, ζάχαρη και η άλλη που χρησιμοποιείται έμεσα η ζάχαρη. Τώρα για το ζαχαροκάλαμο στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ πριν ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα ε, κάναμε τεράστιες εισαγωγέ από τις χώρες ΑΚΕ. Θεωρούσαμε ότι ήταν μια υποχρέωση για μας. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα έχουμε τους ε, ε, επεξεργαστές ε, ζαχαρόδοθλου. Μπορούν να πάρουν τεράστιες ποσότητες, όμως για το ζαχαροκάλαμο είναι διαφορετικά τα πράγματα και υπάρχουν σημαντικέ δυσκολίε. Ο πως ποτέ δεν νομίζω ότι αντιμετώπισε το ζήτημα. Και τέλο. για την υγεία υπάρχει μία εκστρατεία κατά τη ζάχαρη αυτή τη στιγμή, γιατί λένε ότι είναι ανθυγινή. Όμω, διάβασα χθε ε, στις ε, εφημερίδες ότι πρέπει να, διαβάζουμε, να καταναλώνουμε περισσότερη σοκολάτα ε, για να προστατεύσουμε την υγεία μα, περιλαμβάνει όμως ζάχαρη. Ποια είναι λοιπόν η υγιεινή και ανθυγιεινή επιλογή. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σα γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαζό, το βασικό ζήτημα είναι η κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης ε, και γλυκόζης το 2017 με μεγάλες προεκτάσεις για τον ανταγωνισμό και πτώση των δημών. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε ότι υπάρξει πολύ ισχυρότερο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών που παράγουν ε, αλλά να δούμε και τι συμβαίνει παγκοσμίω, ποια είναι η τάση. Ο ανταγωνισμό ε, στο πλαίσιο τη Τίτη, για παράδειγμα, με ε, την αντίστοιχη αγορά τη Αμερική. Θα είναι πολύ σημαντικέ οι προεκτάσει. Νομίζω ότι ε, πρέπει να περιμένουμε και τι αποφάσει τη Βραζιλία και τη ΗΠΑ για τα βιοκαύσιμα. Η Γαλλία είναι το μοναδικό κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει ε, ζαχαροκάλαμο, που είναι κρίσιμη σημασία κλάδο, ιδίω για τι υπερπόντιες περιοχές μας που πρέπει να προστατεύσουμε. Παρότι είναι μικρή η παραγωγή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πρέπει να τις προστατεύσουμε. Επίση, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τι υποχωρήσει αυτέ τι διαπραγματεύσει για να μην αποσταθεροποιήσει την αγορά και ε, να διατηρηθεί η τελωνική δεσμολογική προστασία. Νομίζω ότι η Γαλλία θα συνεχίσει και θα επιδιώξει την διαφοροποίηση της ε, παραγωγής και την έρευνα ε, στον τομέα αυτόν. Ξέρετε ότι και ο γαλλικός κλάδος έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Κύριος Γιάρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν επεκτάθηκε η κοινή αγορά ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δόθηκε η δυνατότητα σε περισσότερους παράγοντες να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, όπως μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα το οποίο χαροποίησε ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, η οποία μας είπε ότι όντως γίναμε τελικά πιο ανταγωνιστικοί ως κλάδο ζάχαρης, αλλά βλέπουμε, συζητώντας για τον κλάδο αυτό, ότι ενδεχομένως τα πράγματα να μην είναι τόσο θετικά, γιατί ε, αν χάσουμε τελικά την κοινή οργάνωση αγοράς ε, για τον τομέα αυτόν, τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε και τις τιμές, οι οποίες όπως είδαμε αυτή τη στιγμή καταραίουν. Και βλέπουμε ότι χώρες όπως η Βραζιλία ετοιμάζονται για την περίοδο μετά το 2020, όπου υποτίθεται ότι θα έχουμε ακόμα πιο χαμηλές τιμές, οι οποίες θα βάλουν κατά τελικά του κλάδου ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε λοιπόν για έναν πολύ σκληρό ανταγωνισμό που μας περιμένει όσον αφορά τα προϊόντα αυτά. Θα είμαστε πραγματικά εμεί σε θέση να συμμετέχουμε στην παγκόσμια αγορά χωρίς να μειώσουμε περαιτέρω τις τιμές μας. Πραγματικά αμφιβάλλω. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Αν όχι, να σας υπενθυμίσω την συζήτηση που είχαμε για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να επανέλθουμε στα έγγραφα αυτά που είχαμε χρησιμοποιήσει τότε. Ακόμα και δεν θυμάστε εσείς τι συζητούσαμε τότε, τουλάχιστον ε, θυμούνται όλα αυτά τα ζητήματα οι καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν, να δούμε ποιες μεταρρυθμίσεις εγκρίναμε παλιότερα και ποια λάθη κάναμε, πού σφάλαμε. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εμπλουτίσει λίγο τη συζήτηση, τα όσα είχαμε πει στο παρελθόν στους παραγωγούς ζαχαροτέφλων. Να ζητήσω τώρα από τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να απαντήσει σε ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω μου δίνετε τη δυνατότητα να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα. Πρώτον, η υφιστάμενη κατάσταση την οποία δεν είχαμε προβλέψει και η οποία έχει προκύψει από το γεγονός ότι συσσωρεύτηκε τεράστια ποσότητα ζάχαρης η οποία θα μεταφερθεί στις ποσοστώσεις της επόμενης περίοδου και η α, σημαντικότατη μείωση των τιμών. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε καταπληκτικά έτη όσον αφορά την παραγωγή της ζάχαρης. Είχαμε μία η οποία ξεπερνούσε τα 700 ευρώ τον τόνο. Αυτό συμβαίνει πάντα στον τομέα της γεωργίας. Ξέρετε ότι μπορεί να έχουμε δύο-τρία καλά χρόνια, ξαφνικά ένα κακό έτος και έπειτα να ακολουθήσει μια καλή χρονιά και το καθεξής. Αυτή τη διακύμανση παρουσιάζει συχνά η παραγωγή στον τομέα της γεωργίας ανεξάρτητα από τον κλάδο. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να εμένετε μόνο σε αυτή την κακή χρονιά που είχαμε ή να είστε τελικά απεσιόδοξοι, γιατί ξέρετε ότι μιλάμε για μια κακή χρονιά η οποία ακολουθεί μετά από δύο-τρία πολύ καλά χρόνια και μάλιστα δύο εξαιρετικά καλά χρόνια. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να αντιδράσουμε στην εφιστάμενη κατάσταση. Τα εφιστάμενα μέσα δεν μας επιτρέπουν να αντιδράσουμε σωστά. Για παράδειγμα, αυτή ε, η ιδιωτική αποθήκευση. Οι συνθήκες ε, που προβλέπονται στον κανονισμό δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το μέσο. Το να περιορίσουμε από την άλλη τις εισαγωγές. Μα καταλαβαίνετε ότι είναι η τιμή της ζάχαρης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τελικά αποθαρρύνει τις ε, εισαγωγές. Και για να απαντήσω στον κύριο Νταντάν, οι δικές μας εισαγωγές είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με τα προηγούμενα, τα παρελθόντα έτη, τα δύο τελευταία έτη. Για παράδειγμα, οι εισαγωγές που προέρχονται από τις πιο φτωχές χώρες, από τις χώρες ΑΚΕ, έχουν μειωθεί κατά 200.000 τόνους. 12% η μείωση όσον αφορά τις ε, ποσοστώσεις ε, ΣΥΞΕΛ, αυτές είναι μηδενικές, ενώ θα έπρεπε να είχαμε 650.000 τόνους. 650.000 τόνους αστικά δεν πήραν τη μορφή εισαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική μείωση των εισαγωγών και αυτό είναι απόλυτα λογικό. Οι τιμές αυτές δεν οδηγούν σε περισσότερες εισαγωγές και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν αυξηθεί και εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο και στο κόστος παραγωγής Ξέρετε ότι ο φόρος από την παραγωγή ζάχαρης περνάει στον κοινοτικό προπολογισμό. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι έχουμε ένα κάποιο απόθεμα. Τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά έχουν ήδη περάσει, έχουν ήδη κοστολογηθεί στον κοινοτικό προπολογισμό. Αν ήταν να χρησιμοποιήσουμε ένα απόθεμα θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να τα πάρουμε από κάποιον άλλο κλάδο και δεν έχουμε νομική βάση για να κάνουμε κάτι τέτοιο μια τέτοια μεταφορά κονδυλίων. Κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, ε, μίλησε υπέρ της παραγωγής των ε, πιο απομακρυσμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπερπόντιων εδαφών. Μα γνωρίζουμε πολύ καλά πώς έχει κατάσταση. Είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την παραγωγή από τις ε, περιοχές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά μιλάμε για πολύ εξειδικευμένη παραγωγή ζάχαρης, την οποία όμως την προστατεύουμε ιδιαίτερα κάθε φορά που συνάπτουμε διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εξαιρέσουμε από κάθε διαπραγμάτευση αυτή την εξειδικευμένη μικρή παραγωγή ζάχαρης. Και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό, γιατί ουσιαστικά αντιστοιχεί ουσιαστικά στη βάση της κοινή οργάνωσης αγοράς ζάχαρης μετά το 2013. Αναφέρομαι εδώ πέρα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ενίσχυση ορισμένων τομέων παραγωγής, όχι αναγκαστικά της ζάχαρης, γιατί αυτό ήδη υπήρχε στο παρελθόν, αλλά αναφέρομαι στην ενίσχυση της παραγωγής κάποιων άλλων προϊόντων και την ενίσχυση των καλλιεργητών για τα προϊόντα αυτά, είναι σαφές ότι μιλάμε εδώ για γεωργικά δικαιώματα, για αγροτικά δικαιώματα, τα οποία εφόσον πρέπει να ερμηνευθούν, θα πρέπει αυτό να γίνει από τις γεωργικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ξέρετε πολύ καλά ότι ε, όσον αφορά την ερμηνεία των κοινωτικών διατάξεων αρμόδιο είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, ε, αν έπρεπε εμεί να δώσουμε μία ερμηνεία, θα έπρεπε να ερμηνεύσουμε τι διατάξει τη γεωργική νομοθεσία τη Ένωση, άρα αυτό θα, θα γινόταν από τι δικέ μα υπηρεσίε, από τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ξέρετε ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού ισχύει για όλου και για τα πάντα και επομένω. Είναι λογικό ορισμένοι να ζητούν να δουν αν όντω εφαρμόζεται σωστά το δίκαιο ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν γέννη πάντως μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες, είτε πρόκειται για το TTIP ή για άλλες εμπορικές συμφωνίες, η άποψή μας είναι ότι ο κλάδος της ζάχαρης είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος κλάδος και συνεπώς οφείλουμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τον ευαίσθητο αυτό κλάδο. Ιδίω, όταν καλούμεθα να διαπραγματευτούμε με χώρες οι οποίες ακολουθούν μια ιδιαίτερα προστατευτική πολιτική, ενθαρρυντική πολιτική όσον αφορά τον κλάδο της ζάχαρης. Όταν λοιπόν διαπραγματευόμαστε με τέτοιες χώρες, τότε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις επιδοτήσεις. Καταλαβαίνετε ότι ένας τόνος επιδοτούμενης ζάχαρης δεν αντιστοιχεί καθόλου σε ένα τόνο μη επιδοτούμενης ζάχαρης. Αυτό λοιπόν το επενθυμίζουμε πάντα και μένουμε σε αυτό στα πλαίσια διαπραγματεύσεων. Εγώ πάντως δεν ανησυχώ ούτε γι' αυτό και ούτε ανησυχώ για τα όσα είπαμε για τις ε, χώρες εκείνες οι οποίες ε, επιδοτούν ε, ή θα προστάτευαν ιδιαίτερα τον κλάδο της ζάχαρης. Κάποιος αναφέρθηκε στην Ινδία. Με εκεί πέρα η κατάσταση είναι καταστροφική όσον αφορά τους καλλιεργητές ε, ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται καν. Έχουμε χιλιάδες χιλιάδων ρούπι που οφείλονται στους ανθρώπους αυτούς πρέπει να καταβληθούν ακόμα ως πληρωμές αυτούς τους ανθρώπους και πρόκειται για λογαριασμούς που δεν έχουν καν εξοφληθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για ισχυρή παραγωγή όταν οι ίδιοι παραγωγοί δεν πληρώνονται καν για την εργασία τους. Οι χώρες λοιπόν αυτές έχουν τα δικά τους εγχώρια προβλήματα και ενδεχομένω αυτά να εξηγούν κάπως και την πολιτική που ακολουθούν, που πολλές φορές δεν συνάδει με τη δική μας την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές δεν είναι συμβατή καν με τους κανόνες του ΠΟΕ. Οι επιπτώσεις πάντως από την πολιτική αυτή δεν είναι τόσο επιζήμιες γιατί έχουν τόσα πολλά προβλήματα σε εθνικό επίπεδο αυτές οι χώρες που δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ανησυχούμε για την πολιτική την οποία ακολουθούν και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει η πολιτική αυτή σε εμά. Τώρα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου ζάχαρης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητά μας βασίζεται σε τρεις ενιστώσεις. Πρώτον, το παραγωγικό κέρδος του καλλιεργητή ζαχαρότευτλου. Τα ζαχαρότευτλα είναι όλο και πιο ε, αποδοτικά, παράγουμε όλο και περισσότερη ζάχαρη με μικρότερες καλλιέργειες ζαχαροτεύτλων. Καταφέρνουμε και έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης, η οποία παράγεται από την ίδια τη μικρότερη καλλιεργήσιμη έκταση. Δεύτερη συνιστόσα είναι η αναδιάρθρωση του κλάδου αυτού οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί. Γίνουν επίσης πολύ σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες είχαν πολύ σημαντική απόδοση. Αναφερθήκαμε επίσης στην ε, περίοδο μεταποίησης του ζαχαρότευτλου σε ζάχαρη, η οποία επιμικίνεται και η οποία μπορεί να μην είναι πολύ περισσότεροι μήνες τελικά, αλλά απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο συνολικά. Και το ίδιο ισχύει ακόμα και για τους υπεύθυνου για το ραφινάρισμα της ζάχαρης, οι οποίοι επενδύσαν σε νέα εργοστάσια, σε νέους εξοπλισμούς, οι οποίοι είναι πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί, όπως σας είπα βρίσκονται κυρίως στις περιφερειακές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που δεν υπάρχουν ζαχαρότευτλα και δεδομένου του πόσο σύγχρονες είναι οι υποδομές που χρησιμοποιούν μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό που προέρχεται από τις άλλες χώρες. Αναφερθήκαμε στη Βραζιλία, πολύ σημαντική χώρα για την παραγωγή ζάχαρης, αλλά τι παραπάνω τελικά μπορεί να κάνει η Βραζιλία. Ξέρετε ότι υποτιμάται συνεχώς το νόμισμα της χώρας. Συνεχής υποτίμηση τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Ε, Αυτό είναι ο λεγόμενος πόλεμος των τιμών. Η τρίτη συνιστόσα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ζάχαρη έχει να κάνει με την ίδια την αξία του ευρώ. Η φυστάμενη τιμή του ευρώ, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ καθιστά τον κλάδο της ζάχαρης πιο ανταγωνιστικό. Η απόδειξη είναι ότι καταφέραμε να αυξήσουμε πάρα πολύ σημαντικά τις εξαγωγές μας στα πλαίσια των ποσοστώσεων ζάχαρης. Η ζάχαρη δηλαδή η οποία έγκυται στην τιμή στήριξης προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ποσόστοση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς μιλάμε για, μια, για έναν κλάδο ο οποίος είναι πραγματικά ανταγωνιστικός, αναφερόμαστε σε έναν κλάδο ο οποίος όντως έχει βελτιωθεί και είμαι πεπισμένο ότι αυτή η απαραγωγικότητα, η επιπλέον που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε, πρόκειται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Σίγουρα η κερδοφορία του κλάδου των ζαχαρότευτλων δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Έχουν γίνει σημαντικότερε επενδύσει οι οποίε πρόκειται να αποδώσουν στο μέλλον. Έχουν γίνει πολύ σημαντικέ επενδύσει σε όλο αυτό το τομέα τη ζάχαρη. Βλέπουμε ότι η έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γίνονται επενδύσει, καταλήγουμε σε συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα. Η θετική αυτή τάση δεν πρόκειται να σταματήσει. Και ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο όντω μπορεί να είναι αρνητικό, δεν το ανέφερα, η εθανόλη, η βιοεθανόλη. Προφανώς ξέρετε ότι δεν είναι ευνοϊκή κατάσταση για τη βιοεθανόλη, διότι είναι πολύ χαμηλές οι τιμές των ορυκτών καυσίμων σε σχέση με τις παλαιότερες ιστορικές τους τιμές και από την άλλη η βιοεθανόλη ξέρετε ότι εξάρτηται πάρα πολύ από τους κανονισμούς που έχουμε σε σχέση με την ενσωμάτωση του προϊόντος αυτού στα συμβατικά καύσιμα. Και αυτό, οι κανονισμοί αυτοί πειράζουν αρνητικά αυτή τη στιγμή τον όλο κλάδο. Συνοπτικά λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, προφανώς μπορούμε να πούμε ότι η υφιστάμενη χρονιά, η τρέχουσα χρονιά είναι αρνητική, αλλά έρχεται μετά από δύο-τρία πολύ καλά χρόνια. Δεύτερον, ο ίδιος ο κλάδος έχει καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες και έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και ειλικρινά δεν ανησυχώ καθόλου και τον κλάδο του ραφιναρίσματος, ο οποίος θα έχει πολύ καλή πρόσβαση στην παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από τις χώρες ΑΚΕ και τις πιο φτωχές χώρες χωρίς ποσοστώσεις και μάλιστα θα χρησιμοποιήσει συνεχώς όλο και πιο αποδοτικά όλο και πιο αποδοτικό μοντέρνο εξοπλισμό. Και γι' αυτό το λόγο εν γέννη θεωρώ ότι ο κλάδος της ζάχαρης θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες που θα του προσφέρει στο μέλλον η παγκόσμια αγορά και κυρίως από το 2017 και μετά. Χρονιά κατά την οποία δεν θα υπάρχουν πλέον συγκεκριμένες ποσοστός και περιορισμοί όσον αφορά τις εξαγωγές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Βαίνουμε προς ε, κλείσιμο του σημείου αυτού της μεσής διατάξεως. Δεν ξέρω κατά πόσον εφωτίστηκα για τα θέματα της Ζαχαρέως, λέει ο Πρόεδρος αλλά ας ελπίσουμε ότι θα δούμε καλύτερες ημέρες σχετικά με το θέμα αυτό. Είχαμε κάνει μια μετακίνηση στην ημεσία διάταξη προς τον Ιούλιο. Ε, θα σας ζητούσα τώρα να εγκρίνετε τις ε, συστάσεις των συντονιστών. Το είχατε λάβει και έντυπα και ηλεκτρονικά αυτό από ό,τι αντελήφθην δεν είχαμε σχόλια επ' αυτού και εις ό,τι αφορά στα διάφορα απλώς να πω προς την Κομισιόν για την οδηγία 76-62 σχετικά με το περιεχόμενο οξέως ή τα λύπη και στην 320 κάθε 206 αν ακούσαμε καλά ε, οι συντονιστές τον Μάιο αποφάσισαν ότι η πρόταση αυτή της Κομισιόν πρέπει επί τη βάση του άρθρου 52 να εγκριθεί χωρίς τροπολογίες. Ε, αυτήν την πρόταση θα ήθελα να διαβιβάσω και καθότι είναι υψηλά τεχνικός το θέμα θα το παρουσιάσουμε αυτό στη συνεδρία του Ιουλίου η οποία, καλά νέα, είναι η τελευταία πριν τις διακοπές. 15 και 16 Ιουλίου θα είναι. Έχουμε κάτι άλλο υπό τα διάφορα, κάποια άλλη ερώτηση, οτιδήποτε άλλο, τότε κηρύττω το πέρας της συνεδριάσεως ευχαριστώντας άπαντες για τη συμμετοχή τους.